Έχουμε το ψήφισμα για τη Ρωσία. και ιδίω τις περιπτώσει Έρστον Κόβερ και Όλεξ Σέντσοφ Αλεξάνδρ Κολτσένκο. Ο κύριο Μπρόκ νομίζω ότι έχει να κάνει μια αναγγελία. Α, για το Αζερβαϊτζάν ήταν, με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 3 με ανάταση της χειρός. Υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 και 2 διανατάσεως της χειρός υπέρ. Κατά. Άποχες. Αρχίζει η ψηφοφορία, επαληθεύουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ψηφοφορία του ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Στο επόμενο θέμα. Αγγόλα. Ονομαστική ψηφοφορία, όπως έχει ζητηθεί, αρχίζει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Στο επόμενο θέμα, ψήφισμα για το Αζερβαϊτζάν όπου ο κύριος Μπρόκ από ό,τι μου είπαν θέλει να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, Ελπίζω να μην αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να ασκηθεί σοβαρή κριτική κατά του Αζερβαϊτζάν για τις παραβιάσεις των εθνικών δικαιωμάτων. Σοβαρή κριτική. Και γι' αυτό μου φαίνεται πολύ καλό το ψήφισμα. Από την άλλη όμως πλευρά δεν μπορούν τα ψηφίσματα, τα κατεπήγοντα μάλλον, να μετατρέπονται σε έναν τρόπο να ε, διατυπώνουμε πολιτικές θέσεις χωρίς ε, προηγούμενη συζήτηση με επιτροπές και επικύρωση των θέσεων και χωρίς συμφωνία για το αν θα πρέπει να υπάρχει η νότια γραμμή ε, προμήθειας ενέργειας ε, και αν θα πρέπει να εξαρτώμαστε μόνο από τη Ρωσία. Χρειάζεται μια λογική συζήτηση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές. Και γι' αυτό σας καλώ να λάβετε υπόψη τη θέση αυτή για να πούμε ότι μπορεί να βγει αυτή η γραμμή, αυτά τα σημεία, τα επίμαχα από το ψήφισμα. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε με ψηφίσματα τα οποία συζητιούνται την Τετάρτη και ψηφίζονται την Πέμπτη ή καθορίστε το κείμενό του Τετάρτη και συζητούνται και ψηφίζονται την Πέμπτη να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε διαπραγματεύσει με την Κίνα, Φερρυπίνη ή όχι ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να είμαστε λογικοί και να βγει το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη. Deci, domnul Broc a făcut sugestia... Κύριε Μπροκ, Προτείνεται δηλαδή μία τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ τους συναδέλφους, το εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να μας επισημάνουν εάν είναι υπέρ μιας τέτοιας προτάσεως. Κύριος Παντσέρη. Ειλικρινά κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα την πρόταση. Αν αυτή ήταν ε, το να διαγραφούν ορισμένα σημεία από το ψήφισμα ή αν αφορούσε κάτι άλλο. Αν ε, πρόκειται για διαγραφή, εντάξει, υπάρχει ελευθερία ψήφου εννοείται. για το κείμενο που όλοι λάβαμε. Αν όμως πρόκειται για αναβολή της ψηφοφορίας ε, όσον μας αφορά, εμείς θέλουμε να παραμείνει η ψηφοφορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν, γιατί πιστεύουμε πως αυτό το κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να εκφραστεί. Τώρα βέβαια το σώμα είναι κυρίαρχο. Καλώς. Εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Μπροκ ζητάει τροποποίηση της ημερησίας διατάξεως. Γι' αυτό και ρωτώ τις πολιτικές ομάδες εάν τη δέχονται την τροποποίηση αυτή. Κυρία τσέκει έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αλλά έχω να πω τα εξή δύο πράγματα. Αφενός, από ό,τι εγώ γνωρίζω, δεν είναι δυνατόν σε τέτοια φάση διαδικασίας να αλλάζει η ημερήσια διάταξη. Το έχουν επισημάνει οι ε, υπηρεσίες μας και στο παρελθόν. Από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να ανεβληθεί η ψηφοφορία του ΕΛΚ. Και δεύτερον, το ΕΛΚ ήταν και εκείνο μέσα στις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να ζητήσει, σε, ε, ζητήσει χωρίς τη ψήφο, σε τμήματα ψηφοφορίας για ορισμένα σημεία. Προφορικές τροπολογίες ζητήστε αν θέλετε, αλλά όχι και αναβολή της ψηφοφορίας. Εμείς είμαστε κατά και της αναβολής ψηφοφορίας και τη διαγραφή σημείων του κειμένου που θα ήταν δυνατό ούτω ή άλλω από ό,τι γνωρίζουμε τον κανονισμό μέσω των προφορικών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρόκ. Πρόεδρε, ας αποφασίσει το κοινοβούλιο. Το πιο απλό είναι αυτό. Ας αποφασίσει το σώμα. Η συζήτηση έγινε, δεν αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη. Είναι καθιερωμένο σαν πρακτική στο κοινοβούλιο. Κάποιες φορές να μην γίνεται η ψηφοφορία, να βάλετε η ψηφοφορία. Δεν με βοηθάει, νομίζω, δεν είναι χρήσιμη η τεχνητή αυτή η ερμηνεία του ε, κανονισμού. Σε 14 μέρες, 15 μέρες το συζητάμε, το ξαναφέρνουμε. Στο Στρασβούργο, στη Μήνη, στο, στη Μήνη του Σεπτεμβρίου, αν θέλετε πιο νωρίς. Το απλούστερο είναι αυτό. Για να βρούμε μεταξύ μας μία λύση. Και έτσι να εξασφαλίσουμε ευρύτατη υποστήριξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Για την καταδίκη δηλαδή των παραβιάσεων δεν μας αλλάζει τίποτα για τις 5-10 ε, μέρες. Αλλά φανταστείτε τι ζημιά μπορεί να προκληθεί εάν δεν περάσει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε να μας λέτε «Α, δεν μπόρεσατε να συμφωνήσετε και άρα κρίμα για σας». Πρόεδρος, κοιτάξτε με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε οι περιπτώσεις είναι δύο. Είτε βγαίνει το θέμα από την ημερήσια διάταξη Α, δεν είναι δυνατό. Πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατό δυνάμει του κανονισμού γιατί είμαστε στα κατεπήγοντα. Δεύτερον, τροποποιείται η ημερήσια διάταξη. Εγώ τηρώ αυστηρά τον κανονισμό των εργασιών. Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση θα ήταν να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη εάν και μόνο εάν το δεχθούν όλες άπασες οι πολιτικές ομάδες. Μία ήδη έχει δηλώσει ότι δεν το δέχεται. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Παρακαλώ, κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα, το θέμα διαδικαστικά είναι απλό, γιατί οι συνάδελφοι δεν ήταν στη συζήτηση. Ο κύριος Πρέντα, ο οποίος είναι και από αυτούς που έχει καταθέσει το ψήφισμα, είπε ότι το ΕΠΠ θα ζητήσει αναβολή της ψηφοφορίας αυτή είναι και το νόημα. βάλτε το στην ψηφοφορία για το αν θα αναβάλουμε την ψήφιση του ψηφίσματος ναι ή όχι. είναι πολύ απλό. Ε, Έχω ακόμα δύο συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Κύριε Βαλενσιάνο. Κύριε Βαρόγκ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δώσαμε το λόγο σε ορισμένους συναδέλφους, θα δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τα κατεπήγοντα τίθενται σε ψηφοφορία μετά το πέρας της συζήτησης. Όποτε δεν δεχθεί να ε, ε, συμμετάσχει ε, σε μια λογική διαπραγμάτευση το ΕΛΚ και να χάσει, αυτό κάνει. Έτσι και αυτή τη φορά. Σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε. Έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα για το Αζερβαϊτζάν. Ο κύριος Κοράο έχει στήσει το λόγο. Εγώ που θέλω να απαντήσω στον κύριο Μπρόκ, γιατί λέει πως δεν ε, πρέπει να το κάνουμε ζήτημα κανονισμού, αλλά πολιτικό ε, ζήτημα. Εγώ θεωρώ πως είναι παράλογο να μπορεί κάποιος να πει πως ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί στην ε, Επιτροπή και όχι ε, στην Επιτροπή όπως για το Αζερβαϊτζάν, ενώ για αυτό που κάναμε για τη Ρωσία, Ρωσία ήταν εντάξει. Δεν μπορούμε να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Στο Αζερβαϊτζάν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Έχουμε ψήφισμα. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς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 Ε, αναβάλλονται ψηφοφορίες για ψηφίσματα που έχουν ζητηθεί και κατευθεί. Εάν λοιπόν ισχύει αυτό και το επιβεβαιώνουν και οι υπηρεσίες, δεν επιτρέπεται καν να συζητείτε το αίτημα του κυρίου Μπροκ. Και αυτό το επισημάνατε εσεί, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε να σας πω λέει ο Πρόεδρος. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε. Και ο μόνος τρόπος να ψηφίσουμε θα ήταν να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη. Για να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη θα έπρεπε να υποστηρίζουν το αίτημα όλες οι πολιτικές ομάδες. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει και άρα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Σημείο 7. Αδιανατάσσεως ισχυρός. Το σημείο 7. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. It's no manipulation, Mr. Δεν υπάρχει καμία χειραγώγηση ή χειρισμός εδώ. Ακριβώς έτσι είναι γραμμένο. Για να το επαναλάβω. Για μια ακόμη φορά περνάμε στην ψηφοφορία για την παράγραφο 7 πρώτο τμήμα. Υπέρ, παρακαλώ, σκώστε τα χέρια. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του ΣΥΜΕΠΤΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 διανατάσσω στις χειρός ψήφι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Este închis. ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η τροπολογία 2. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο τώρα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του αρχικού κειμένου ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18, παράγραφος 18, το αρχικό κείμενο, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι ΠΕΡ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Από την κυρία Σχάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας απασχολήσω. Μια διόρθωση μόνο για την αποστολή οντί για τις ε, παρατήρηση εκλογών. Ε, η τελευταία πρόταση της παραγράφου ζητούμε να διαγραφεί από το Asian Observation μέχρι Electoral Environment. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος που είναι αντίθετος προς την τροπολογία. Αν όχι, περνάμε σε ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίζουμε το σημείο αυτό όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη. ΕΜ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχέδιου ψηφίσματος. Περ, Κατά αποχές θα προτιμήσω να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Τροπολογία 6, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία και τα δύο άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημείο 6. Τρία τμήματα ονομαστικά και τα τρία, άρχεται η ψηφοφορία το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 7. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα παράγραφος 9 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Τώρα ψηφίζουμε ονομαστικά την παράγραφο 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε μια προφορική τροπολογία από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ για το 11. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. πολύ απλή τροπολογία για την παράγραφο 11 στο τέλος ε, να προσθέσουμε taking into account the best interest of the child, λαμβάνοντας υπόψη ε, τα συμφέροντα του παιδιού. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος που είναι αντίθετος με την τροπολογία αυτή, με την προφορική αυτή τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν με την τροποποίηση. Ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Παράγραφος 11 λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να κυρωθεί ψηφοφορία. Deci, încă o dată, încă o dată să fie toată lumea pe aceeași lungime de undă. Για να είναι σαφές για όλους, ψηφίζουμε την παράγραφο 11, λέει ο πρόεδρο όπω τροποποιήθηκε μετά από την πρόταση τη κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κυρία Κοράτσα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μιλάμε για την τροπολογία 11. Ψηφίζουμε την παράγραφο 11, επί της οποίας προστίθεται η προφορική τροπολογία. Να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των παιδιών. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω όλη την παράγραφο cred că lumea știe despre ce este vorba. Νομίζω γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι το περιεχόμενο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την παράγραφο 11 όπως τροποποιήθηκε από την προφορική τροπολογία της κυρίας Κοράτσα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Adoptat. Adoptat. Εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Τροπολογία 11 στην παράγραφο 12. I am told that the interpreters might have got it wrong. Ίσως υπήρξε κάποια παρανόηση. Μάλλον από τη διερμηνία. Μιλάμε για την τροπολογία 11 στην παράγραφο 12, ονομαστική ψηφοφορία. Ίσως κάπου έγινε κάποιο λάθος σε κάποιες γλώσσες. Λοιπόν, πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 τώρα. Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένα, Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. εγκρίνεται. Απολογιατρία υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 15, το αρχικό κείμενο δηλαδή, σε δύο τμήματα. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Αιτιολογική σκέψη J. Αρχικό κείμενο δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Διαντάσεως. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Εποχές, Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο τώρα του σχεδίου ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία, τώρα περνάμε στο ψήφισμα που αφορά τη Μέση Ανατολή. Αναδιαδικαστικό. Ζητώ συγγνώμη σε αυτή την τελευταία, για αυτή την τελική παρέμβαση. Υπήρξαμε, προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε. Θα ήθελα να ε, ζητήσω αν μπορεί να γίνει μια προφορική τροπολογία ε, ε, συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία, γιατί η πρώτη τροπολογία από το ECR είναι επικίνδυνη. Πρόκειται για εθνική κάθαρση και θέλω να θυμίσω ότι το 20% των, πολιτών του Ισραήλ είναι, δεν είναι πολίτες του Ισραήλ και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Αν μπορούμε να κάνουμε ονομαστική κλίση, τουλάχιστον θα πρέπει να βλάψουμε τη, φήμη αυτού του κοινοβουλίου και θα πρέπει να το καταψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Από την πολιτική άποψη κατανοώ αυτό που λέτε. Ωστόσο, αυτό που δεν καταλαβαίνω δεδομένου ότι υπάρχει κανονισμός, είναι ότι έρχεστε τελευταία στιγμή με αυτή την πρόταση, που δεν μπορώ να δεχτώ. Είναι ξεκάθαρο το θέμα λοιπόν. Και προχωράμε στη ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Μάλιστα, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Σημείο 6 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα με διανατάσεως. Ποιοι είναι υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική κλίση για το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία τη ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Avem situația din Belarus. Περνάμε τώρα στην κατάσταση στη Λευκορωσία. Σημείο 6 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Διανατάσσεως της χειρός πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ονομαστική κλίση για την τροπολογία 1 άρχεται πέρας απορρίπτεται Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Διανατάσεως, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωράμε στην ψηφοφορία για την έκθεση Λόπεθ Φοντανιέ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ενέργειας. Παράγραφος 19 αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα διανατάσεως. Πρώτο τμήμα υπέρ. Δεύτερο, ε, κατά, με συγχωρείτε, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 20 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα διανατάσεως. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 σε δύο τμήματα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 44 σε δύο τμήματα, ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 50 ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 51 ονομαστική κλίση άρχεται πέρας εγκρίνεται εκτιμώντας M σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος τώρα, με ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση, έκθεση Ντλαμπαγιόβα, δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 21ο αιώνα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Πέρας. απορρίπτεται. Παράγραφος 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Εγκρίνεται. Ε, αρχικό κείμενο πριν το σημείο 3. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφο 9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διανοτάσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13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 ε, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Δεκαεννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το 19 πάλι για το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ, ε, σε δύο τμήματα ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εντάξει ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται Πέρασε. Απορρίπτεται. Πενήντα Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, τέλος, εγκρίνεται. 71 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 71, ε, ονομαστική κλίση, Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. 73 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασες τη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 74-2 τμήματα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 81 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές και επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84 σε δύο τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 86 τρία τμήματα ονομαστικά. αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 90 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 δύο τμήματα στο πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 101 ονομαστικά, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 102 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 τέσσερα τμήματα ονομαστικά και τα τέσσερα από το πρώτο παρακαλώ αρχής ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται δεύτερο τμήμα έρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη C, λατινικό σε τρία μέρη. Ονομαστική ψηφοφορία και τα τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. F ε, λατινικό σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τελική σκέψη ήταν. Θα κάνουμε επαλήθευση για το F, για το δεύτερο τμήμα του F. Επαλήθευση ηλεκτρονική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη τα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Χρυσόγονου, τρίτη και τεκοστή πρώτη έκθεση όσον αφορά την παρακολούθηση ε, της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείο 5, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. 9. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της 9 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του, μονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και